Pan prezeda. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání je zahájeno. Prvním bodem pořadu jednání je zpráva. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίαση και το πρώτο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης είναι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και χαιρετίζω μεταξύ ημών τον κύριο Φιλίπ Μέιστατ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος θα συμμετάσχει στην σημερινή μας συζήτηση. Θα δώσω όμως καταρχήν για πέντε λεπτά τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση της ΕΤΕ, κάτι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων δραστηριοτήτων της ΕΤΕ. Αν και πρόκειται για μία πάγια διαδικασία, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως κάτι το δεδομένο, γιατί μας δίνει βασικά στοιχεία για το μέλλον της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνα το Δεκέμβριο του 2009 αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί βασικό εταίρο. Κύριε Κούτα, με συγχωρείτε. Θα ήθελα λιγάκι να επιβραδύνετε διότι δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις βελτιώσεις της έκθεσης και θα ήθελα να ευχαριστήσω και το διευθυντικό προσωπικό της ΕΤΕ για την πολύ καλή συνεργασία και τον ε, πρόεδρο Μάιστατ και τον αντιπρόεδρο Κολάτς Άναν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουν αυξηθεί και το χρέος και το έλλειμμα των κρατών μελών. Βλέπουμε όμως ότι παρόλα αυτά μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 θα πρέπει να προβούμε σε μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία και οι τις πάγιες υποδομές. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να το επιλύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΤΕ λοιπόν πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτά τα πλαίσια. Θα λάβω δύο μείζωνα θέματα που απασχόλησαν την ΕΤΕ για την εξυγίαση της οικονομίας. Καταρχήν, τις δανειοδοτήσεις προς τις ΜΜΕ και την προώθηση των προγραμμάτων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΜΜΕ είναι μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μέσα στα πλαίσια της καινοτομίας και της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει στις ΜΜΕ του 2009-2010 χρηματοδοτήσεις 7,5 δις ευρώ. Μέσα στα πλαίσια των μικροεπενδύσεων και μικροχρηματοδοτήσεων φτάσαμε σε 200 εκατομμύρια ευρώ με βάση τις μικροπιστώσεις τα δεδομένα των μικροπιστώσεων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δυσκολίες πρόσβασης στην ΕΤΕ από τους μικροεπιχειρηματίες. Επειδή χρειάζεται λοιπόν ε, καλύτερη διαδικασία ε, επενδύσεων και καλύτερη διαδικασία επιλογής, η ΕΤΕ θα πρέπει να προσδώσει τα διάφορα μέσα στις ε, περιοχές μικροσύγκλησης έτσι ώστε να υπάρχουν δυνατότητες επενδύσεων. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα μικροπρογράμματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και με το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εκδόσεις ομολόγων μέσα στα πλαίσια των ε, δεδομένων που μας προσφέρει το Ταμείο Συνοχής. Επειδή υπάρχει λοιπόν αυτός ο πολλαπλασιωστικός παράγων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα χρήματα για να προωθήσουν τα σχέδιά τους ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία και έρευνα. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν την βιώσιμη ανάπτυξη, τις σιδηροδρομικές ε, διασυνδέσεις, τις οδικές αρτηρίες και τα προγράμματα όπως αυτό του Ναμπούκο για τους αγωγούς φυσικού αερίου. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για το θέμα της διαφάνειας και των φορολογικών παραδείσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η ΕΤΕ να μην συνεργαστεί με μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες των διαφόρων οργανώσεων. Όμως αυτή η κατάλογη δεν είναι ικανοποιητική. Η ΕΤΕ θα πρέπει να προωθήσει την περιοδι... τις περιοδικές υποχρεώσεις αυτών των φορέων. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΕΤΕ συνεισφέρει και στις συνδεδεμένες χώρες ή τις χώρες προς ένταξη για την ανάπτυξή τους. Άρα υποστηρίζουμε τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερο προσωπικό και καλύτερη συμμετοχή των τοπικών φορέων. Κύριε Κούτας, δεν έχετε άλλο χρόνο. Χαίρομαι και θα χαρώ να ακούσω τους παρευρισκόμενους και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο Μίστατ. Στον πρόεδρο της ΕΤΕ. Έχετε το λόγο κύριε Μίστατ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε για άλλη μια φορά και μπορώ σήμερα να συμμετάσχω στην σημερινή συζήτηση που αφορά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούτα, τον εισηγητή, ο οποίος δεν αφιέρωσε τις εργασίες του μόνο στην αναδρομική περιγραφή της τράπεζας, αλλά κάνει και κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Και θα ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτές. Θα ήθελα να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έδωσε μια τρίπλη κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια και καθόρισε τρεις άξονες. Στρατηγική Ευρώπης 2020, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η στήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή κρίση, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, οι απαντήσεις είναι βραχυπρόθεσμες. Και αυτό ισχύει και σε εθνικό επίπεδο, διάσυση των τραπεζών, αλλά και κινητοποίηση της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό σχέδιο το οποίο όρισε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2008 κινητοποίησε με 48 δισεκατομμύρια το 2007 και 78 το 2009 την ευρωπαϊκή οικονομία με νέα λοιπόν κονδύλια, στοχευμένα σε στόχους οι οποίοι θεωρούνται στόχοι προτεραιότητας, ιδιαίτερα για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ανέφερε και ο εισηγητής. Μετά από αυτήν την βραχυπρόθεσμη ε, απάντηση, η οποία μας βοήθησε να ξεπεράσουμε την πρώτη δυσκολία, θα πρέπει να έχουμε και μία πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, Ευρώπη 2020, με πολύ σημαντικούς τομείς, όπως την αύξηση των ε, κινητοποιήσεων στον τομέα της ε, απασχόλησης, την γνώση, την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να συνεισφέρει σημαντικά σε αυτή τη στρατηγική. Το 2010 ήδη χρηματοδότησε με πάνω από 4 δισεκατομμύρια τον τομέα της παιδείας και πάνω από 7 δισεκατομμύρια προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέλει να αυξήσει τα κονδύλια που διαθέτει σε αυτούς τους τομείς, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημιουργώντας εργαλεία χρηματοδότησης κοινά, ιδιαίτερα όσον αφορά την Risk Finance Facility, διότι τέτοια εργαλεία επιτρέπουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό να δράσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μπορούμε δηλαδή να αυξήσουμε τις επενδύσεις με το ίδιο ποσό και την ίδια ώρα αυτό το κοινό εργαλείο χρηματοδότησης μειώνει το βάρος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή με το ίδιο κεφάλαιο μπορεί να χορηγήσει περισσότερα δάνεια. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την δυνατότητα χρηματοδότησης της έρευνας, μπορούμε με 390 δισεκατομμύρια και με 700 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να δώσουμε, να χορηγήσουμε δάνεια για πάνω από 6 δισεκατομμύρια και να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που ξεπερνούν τα 16 δισεκατομμύρια στον τομέα της έρευνας. Είναι λοιπόν προφανέ ότι η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη στιγμή που θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με άλλα θεσμικά όργανα και άλλου ε, χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Δεύτερο άξονα καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο και τι δραματικέ συνέπειέ Αυτό είναι μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, οι συνέπειες αυτού ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη να επενδύσουμε με τρόπο μαζικό στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην τεχνολογία στον τομέα της ενέργειας. Προγράμματα που έχουν σε σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών ξεπερνούν τα 20 δις τουλάχιστον, δηλαδή 30% των συνολικών δανείων που χορηγήσαμε. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 6,2 δις, κυρίως προγράμματα παραγωγής ενέργειας αιωλικής και ηλιακής, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενεργειακής προγράμματα που ξεπερνούν τα 2,3 δις το 2010 και θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια με τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα στα δημόσια κτίρια, αλλά και στις κατοικίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, επενδύσεις που έχουν σαν σκοπό και τη βελτίωση των ε, μέσων μαζικής μεταφοράς, την μείωση των ε, ΙΟΤΑΧΗ που ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια το 2010. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την στήριξη εξοικονόμησης ενέργειας ενεργειακής αποτελεσματικότητας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επεξεργαζόμαστε μια περίπλοκη από τεχνολογικής απόψεως μεθοδολογία με σκοπό να αξιολογήσουμε με ακρίβεια το ίχνος του άνθρακα, το αποτύπωμα του άνθρακα. Ο τρίτος άξονας της πολιτικής μας αφορά την εξωτερική πολιτική, η οποία βεβαίως χρειάζεται οικονομική στήριξη. Αυτό το κατάλαβε και η Κίνα, η οποία στηρίζει τις εξωτερικές της δραστηριότητες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αναπτύξει μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτήν την πολιτική και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και αυτό βεβαίως είναι μία από τις ε, προτάσεις της έκθεσης Κόμτοσού, και βεβαίως εάν το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η τράπεζα θα στήριξει όπως το ορίζουν εξάλλου και οι δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τι τρει κατευθυντήριε γραμμέ τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 2020. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος λοιπόν ο κύριος Σεύκοβιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κούτα για μια εξαιρετική έκθεση και να καλασορίσω εδώ τον πρόεδρο της τράπεζας κύριο Μάιστατ γιατί είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Ολομέλεια να ακούσει και τις απόψεις σας αλλά και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και να ακούσει τα συγχαρητήριά μας για την άμεση απόκριση που έδωσε η ΕΤΕ ε, στην χρηματοπιστωτική κρίση. Έτσι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητα στην αγορά κάτι το οποίο ήταν σημαντικό και για την ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τους υπόλοιπους εταίρους μας στον κόσμο. Κατάφερε η ΕΤΕ να αυξήσει τη δραστηριότητά της και να στοχεύσει τη χρηματοδότηση στους κλάδους οι οποίοι βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η Κομισιόν θα συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο. Στήριξη της πολιτικής συνοχής και μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αποτελούν τους στόχους μας για το μέλλον. Εμείς με την ομάδα της ΕΤΕ θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να παράσχουμε τα, κατάλληλα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοδοτικά μέσα κατά της αλλαγής του κλίματος, το Jasper, το Jeremy και το πρόγραμμα το καινούριο το αίμα. Συμφωνούμε με τα όσα είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε όντως περισσότερο ποιοτικά εργαλεία για καλύτερη και μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη βέλτιστη κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα όσα κάνετε εσείς δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια βέλτιστη χρήση του κεφαλαίου που έχετε. Γιατί βέβαια έχουμε κάποιες δράσεις ψηλού κινδύνου που είναι μεγαλύτερης κεφαλαιολογικής ανάλωσης αλλά που δίνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία θεωρούμε πως τα καινοτόμα εργαλεία αν χρησιμοποιηθούν μαζί από ε, ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς όπως η ΕΤΕ θα φέρουν αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν εγγυήσει και ομόλογα τα οποία έχουν καταφέρει όχι μόνο να ηρεμήσουν τις αγορές αλλά να εξασφαλίσουν και κονδύλια από τρίτους και η χρήση των κοινών αυτών εργαλείων και η ανάληψη από κοινού κινδύνου με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης απελευθερώνει κεφάλαια έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει καλύτερα τους ίδιους πόρους η ΕΤΕ. Τελικά αυτό τι σημαίνει. Περισσότερα έργα θα στηριχθούν για την Ευρώπη της 2020 για να εξυπηρετηθεί η σχετική στρατηγική και για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτήν. Η Ευρώπη του 2020 και τα ομόλογα έργων που έχουν δεσμευθεί νομίζω ότι αποτελούν το καλύτερο παράδειγμα και στη στρατηγική αυτή έχουμε ε, κάνει μια έκκληση για μεγάλες επενδύσεις διασυνοριακές έτσι ώστε να έχουμε ευφυεί ευφυείς αναβαθμισμένες και διασυνδεδεμένες υποδομές στα πλαίσια πάντα της Ευρώπης του 2020, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες. Εκεί είναι οι βασικές υποδομές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ε, πιθανή κλάδη που θα μπορούσαν να θέσουν τα θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον. Και χαίρομαι που στηρίζετε εσείς τις πρωτοβουλίες αυτές στην έκθεση τη δική σας. Τώρα, στα πλαίσια της προετοιμασίας των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολιετές πρόγραμμα πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτή τη στιγμή μια στρατηγική ανάλυση των όσων συμβαίνουν για να έχουμε μια βέλτιστη χρήση αυτών των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων έτσι ώστε μαζί με τα όσα κάνει η ΕΤΕ να χρησιμοποιήσουμε την πείρα που έχουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ε, σε επίπεδο αγορά. Για τι εξωτερικέ ενέργειε που αναλαμβάνει η ΕΤΕ και για δράσει χρηματοδότηση εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί στηρίζουμε την αύξηση των οροφών που πρότεινε ε, ε, το Κοινοβούλιο στα πλαίσια τη ενδιάμεση αναθεώρηση, στα πλαίσια του πολιτού προγράμματο. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο προτείνει το αύξηση για την περιοχή τη Μεσογείου μα βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Επίση, η στήριξη της ε, μετάβασης προς μια ε, ε, δημοκρατική κοινωνία των εταίρων μας σε άλλες περιοχές στο Νότο. Χρειάζεται δεν να χρησιμοποιήσουμε και ροές από προηγούμενες επενδύσεις στην περιοχή της Μεσογείου έτσι ώστε να έχουμε και διαθέσιμο κεφάλαιο από ιδιωτικούς επενδυτές high risk στην περιοχή. Αυτές οι επιπλέον ανάγκες που εμφανίζονται σήμερα Χρειάζονται βέβαια περισσότερους πόρους προσωπικό που να είναι εξοικειωμένο με την αναπτυξιακή ε, βοήθεια και χρηματοδότηση. Για την εξωτερική εντολή της ΕΤΕ εμείς θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας για να μελετήσουμε το πώς μπορεί να βρεθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανάπτυξη έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε ε, την χρήση δανείων που παρέχεται και από την ΕΤΕ αλλά και από άλλα πολυμερή ή διμερή όργανα. Τέτοιου είδους πλατφόρμα θα δημιουργήσει συνέργειες και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕ και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν αναφέρομαι στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Ανάπτυξης και Αναδιάρθρωσης και της ΕΤΕ που έχει ήδη υπογραφεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Οντί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε μάλιστα, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που δείχνετε στις προτάσεις μας. Σαν πρόεδρος μιας διακυβερνητικής τράπεζας θα μπορούσατε να μην είστε τόσο ευαίσθητος στις ε, δικές μας σκέψεις. Όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά το κοινοτικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων, θα ήθελα να πω τα εξή. Για την ασφάλεια, είπατε ότι θα θέλατε να είστε ο οικονομικός βραχίωνας της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα τριπλό αλφα βεβαίως σαν αξιολόγηση, θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η πολιτική μας στον τομέα αυτό. Πρέπει να στηριχτούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα μπορούσε την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να στηριχθεί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μία ή περισσότερες ρυθμιστικές αρχές. Περιμένουμε τις προτάσεις σας, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι η πρότασή μας είναι να γίνει μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έτσι ώστε αυτό το διακυβερνητικό όργανο να μπορέσει σιγά σιγά να γίνει κοινοτικό. Ευχαριστούμε. Τώρα, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, η κυρία Χούμπνερ καταρχήν, εξ του ΕΛΚ. Πρόεδρε Μάιστατ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να μιλήσω για το μέλλον πρωτίστως και θα ήθελα να θίξω τρία σημεία, την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της Ευρώπης. Και αυτό σημαίνει επενδύσεις και χρηματοδότηση των επενδύσεων. Το θεμητό ερώτημα είναι από πού θα προέρχεται η χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι η απάντηση, στην απάντηση εγγύεται το μέλλον της Ευρώπης με βάση και τη συνεισφορά της ΕΤΕ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα επόμενα έτη θα υπάρχει παγκόσμιος ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση, περαιτέρω περικοπές και ο τραπεζικός τομέας θα γνωρίζει μεγάλη ανασφάλεια μέσα στα πλαίσια των πάγιων χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. Και βεβαίως ο κοινοτικό προπολισμό θα είναι πολύ περιορισμένος για να μπορέσει να επιλύσει τα προβλήματά μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την κίνησή σας προς καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης και εκτιμούμε τη μέχρι τώρα δραστηριότητά σας, αλλά αυτός ο επιμερισμός ε, κινδύνου δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει αν δεν υπάρχει η αρρωγή και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ένα ίσως καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά πολλές φορές μπορεί να πνίξει τις φιλοδοξίες μας. Γι' αυτό μιλάμε για ένα αριθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα ήταν πιο θαραλέο και θα τονίζει και τη μότχλευση και τον καταλητικό ρόλο της ΕΤΕ, έτσι ώστε να βρεθούν μέτρα αναπερίπτωση. Και ελπίζουμε ότι θα κινηθείτε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ε, μια πλέον θαραλέα ρυθμιστική πολιτική και θα σας υποστηρίξουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Μπέρμαν, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κούτας για την εξαιρετική έκθεση ετήσιων δραστηριοτήτων της ΕΤΕ για το 2009. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για τη σχέση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι από κοινού νομοθέτη σε σχέση με τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕ ως προς τις γείτονες χώρες και τις υποανάπτυξη χώρες. Όμως το Συμβούλιο φαίνεται ολιγορεί ως προς την αναθεώρηση αυτής της εντολής ε, της ΕΤΕ για τις εξωτερικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι η πρότασή μας ε, δεν γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο σε σχέση με τα μέτρα της ΕΤΕ για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών ή της ε, χρηματοδοτήσεις, μικροχρηματοδοτήσεις ιδιαίτερα. Αν αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να ξαναδεί πώς θα ορίσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου. Γιατί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βρίσκονται σε ίση βάση τώρα ως προς την κοινή νομοθέτηση και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες της ΕΤΕ. Θα πρέπει λοιπόν οι δύο κοινοί νομοθέτες να δέχονται ο μεν τον δε, διότι δεν μπορούν να απορρίπτονται οι προτάσεις του Κοινοβουλίου εξορισμού από το Συμβούλιο. Η στάση του Συμβουλίου είναι απαράδεκτη και επίσης είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι σήμερα το Συμβούλιο δεν παρευρίσκεται εδώ η ΕΤΕ αποτελεί έναν βασικό μοχλό δράσης για την εξωτερική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανάπτυξη τρίτων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Χρειάζεται μια δημόσια τράπεζα για όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις αναπτυσσόμενες χώρες βεβαίως. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια όπως ορίζει η συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να προωθήσουμε την καταπολέμηση της ε, φτώχειας για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η κυρία Κουλάρ εξ των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Καλημερίζω ε, τον πρόεδρο τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα ήθελα να σα πω το εξή. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε την έκθεση, μιλήσαμε για την ανάγκη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κάτι το οποίο ήταν επιτακτικό λόγω τη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έδειξε ότι ήταν υπερβολικά κοντόφθαλμη η τακτική που είχαμε ακολουθήσει μέχρι τότε. Δηλαδή, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και εκεί το δικό σα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει πολλά να δώσει. Για τον νότο της Μεσογείου πιστεύω πως ίσως θα πρέπει εμείς να ευαισθητοποιηθούμε για τις ανάγκες που δημιουργούν οι ενεργειακές μας επιλογές. Θα ήθελα πάντως να σας στηρίξω και να σας πω πάντα στο κοινοβούλιο αυτό θα βρείτε ε, βουλευτές να σας στηρίξουν και όπως είπε ο συνάδελφος ο Ντί, είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει να ελέγχουμε καλύτερα μία σειρά από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί προς τα εκεί έχουμε κοιμηθεί, θα πρέπει να δούμε κάποιες καινοτόμες ιδέες. Για παράδειγμα, τα ομόλογα έργων είναι μια καλή πρόταση. Ίσως θα έπρεπε να δούμε και τα σδίτη για παράδειγμα, για να δούμε με ποιο τρόπο έχει οργανωθεί αυτή η συνεργασια δημοσιοδιωτικού κλάδου, να δούμε ποιος θα πρέπει να έχει ε, δικαίωμα συμμετοχή. Είναι ένα εργαλείο χρήσιμο, όπως επίσης και κεφάλαια, όπως το Marguerite που έχουν συσταθεί στην Ευρώπη, που στηρίζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, αλλά θέλουμε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και παρακολούθηση και έλεγχο. Νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας στηρίζουμε και θα θέλαμε όλες αυτές οι τελευταία, όλα τα τελευταία γεγονότα να μας παροτρύνουν να κοιτάξουμε το μέλλον και να το ταινίσουμε βλέποντας το σε όλο το το εύρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κομφέρα, επόμενος από τους Πράσινους. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ξέρετε ότι η πράσινη θεωρεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σαν ένα όργανο στήριξης της δημόσιας πολιτικής. Και ακριβώς επειδή το θεωρούμε πολύ σημαντικό, είμαστε και πολύ απαιτητικοί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μια πραγματική τράπεζα με όλες τις ε, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μιας τράπεζας, το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι ίσως θα έπρεπε να δεχθεί και επιπλέον δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Από την άλλη μεριά όμως πρόκειται για τα χρήματα των ε, Ευρωπαίων φορολογούμενων, άρα θα πρέπει να υιοθετηθούν κανόνες που ξεπερνούν αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Θα ήθελα να επιμείνω παρουσιάζοντας κάποια σημεία στα οποία πιστεύω ότι παρόλη την πρόοδο που έχει γίνει θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειες. Το πρώτο θέμα είναι η φορολογική παράδειση. Είναι μια σημαντική υπόθεση. Η κρίση μας έδειξε ότι συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και το όλο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει να ευαισθητοποιεί περισσότερο από τους φορολογικούς παραδείσους και την ύπαρξή τους. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και για τα δάνεια που χορηγείται στις επιχειρήσεις και τα οποία περνούν από τους φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ξέρω βεβαίω ότι έχετε ε, κάποιες δεσμεύσεις ε, επιχειρηματικού χαρακτήρα, αλλά εάν πραγματικά θέλετε να γίνετε ο βραχίωνας της ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τη χρηματοδότησή σας ζητούμε να θέσετε αυστηρότατους όρους στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν την αλυσίδα των αξιών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα του ΟΣΑ. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Έλεγχος και διακυβέρνηση. Η Σιλβί Γκουλάρ ανέφερε το θέμα αυτό μόλις τώρα. Πιστεύω θα πρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες, τις συλλογικές ευθύνες και οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνονται με το πιο δημοκρατικό τρόπο. Τρίτο σημείο. Το όφελος της δράσης σας. Είστε μία τράπεζα και φυσικά μετράτε την αποτελεσματικότητά σας σε σχέση με το ρίσκο ε, και το κέρδος. Θα πρέπει όμως το κέρδος και το όφελος να μετρούνται και με άλλο τρόπο. Κοινωνική συνοχή, αποτελεσματική δράση σε άλλους τομείς από αυτόν του οικονομικού κέρδους. Και πιστεύω ότι αυτά τα ωφέλη, αυτά τα πλεονεκτήματα εκτός των καθαρά οικονομικών και χρηματοπιστωτικών θα πρέπει να μετρηθούν με έναν τρόπο και θα πρέπει να διευρυθούν, διότι δεν περιορίζονται μόνο σε νομισματικά και χρηματοπιστωτικά μετρήσιμα κέρδη και ωφέλη. Λέει με ρητό τρόπο η έκθεση ότι θα πρέπει να υλοποιήσετε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά 80% το 2050 θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε μονάδες που λειτουργούν με άνθρακα. Κύριε Κομφά. Κύριε Κομφά. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα. Ναι. Πώς δέχεστε τη χρήση της ΕΤΕΟΣ ε, ένα όργανο το οποίο για τη δράση του αυτή θα επιβαρύνει ε, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τον Ευρωπαίο και τον Βρετανό φορολογούμενο. Πολύ απλή είναι η απάντησή μου. Ο Ευρωπαίος φορολογούμενος κοιτά αυτή τη στιγμή τα καθαρά ειδικά συμφέροντά τη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξυπηρετεί πολύ καλύτερα το κοινό συμφέρον από τις ιδιωτικές Βρετανικές τράπεζες. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Σουίνμπερτ εκ μέρους των συντηρητικών. Ευχαριστώ χάσαμε πολύ χρόνο, δαπανίσαμε πολύ χρόνο για τις, μιλώντας για τις χρηματοοικονομικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι υπόλογες. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε, αυτό το, σε αυτή τη νέα εποχή της λογοδοσίας με βάση την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει να λογοδοτούν όλα τα θεσμικά όργανα και η ΕΤΕ, επειδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ΕΤΕ για την χρηματοδότηση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι υπόλογοι. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι η αποτίμηση της δανειοδότησης των δραστηριοτήτων δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται δοκιμές αντοχής και όταν υπάρχει μόχλευση ή κίνδυνος θα πρέπει εξορισμού να ορίζουμε και να λογοδοτούμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το τίμημα το καταβάλουν οι φορολογούμενοι και έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια της ε, δημιουργίας νέων χρηματοπιστωτικών οργάνων. Ευχαριστούμε κυρία Σουινμπέρν, ο κύριος Κλούτε, εξ ονόματος της ΓΟΕ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, κύριε Μάιστρα, τα αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά θα πρέπει με μακροχρόνιο τρόπο να κινητοποιηθούν, να ενισχυθούν οι ενισχύσεις. Αυτό είναι και ο στόχος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Άρα είναι πραγματικά δεσμευμένη στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωση. Περισσότερη διαφάνεια, αηφόρος ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη χρηματοδότηση των στόχων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι αυτά όλα δεν καλύπτονται και αυτό το είπαν πολλοί. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί επικρίνουν συχνά τις διάφορες δραστηριότητες οι οποίες γίνονται χωρίς διαφάνεια όπου τα χρηματοπιστωτικά οι χρηματοπιστωτικέ δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο που καθόλου δεν εξυπηρετεί του στόχου αυτού. Η άποψή μα είναι ότι βεβαίω και θα πρέπει να ακουστούν οι επικρίσεις των μη κυβερνητικών οργανισμών προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότηση βασιζόμενος στα κριτήρια αυτά αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας. Αυτό δεν είναι το μόνο που επικρίνουν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και χρηματοδότηση προγραμμάτων σε τρίτος χώρες που απαιτεί στόχους κοινωνικούς, περιβαλλοντολογικούς και όλα αυτά σήμερα δεν ελέγχονται και δεν μπορούμε να πούμε ανταποκρίνονται στους στόχους Ευρωπαϊκής Ενότητας και στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, τους κοινωνικούς στόχους θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως να τηρούν όλους αυτούς τους στόχους. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η χρηματοδότηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως ιδιαίτερα σήμερα μετά από το ατύχημα, την καταστροφή στην Ιαπωνία. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που δεν είναι πυρηνικές. Θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους, μια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχουμε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Hans Peter Μάρτιν. Την δέχεστε. Ο κύριος Μάρτιν λοιπόν από ό,τι άκουσα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να γίνει ένα εργαλείο, ο να είπατε για την ανάπτυξη. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος. Πώς βλέπετε αυτή την πρόταση παραδείγματο χάρη αυτό που γίνεται σήμερα με τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζας σε τρίτε χώρε στην Κίνα. Ναι, θεωρώ ότι δύσκολο είναι σήμερα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά εκθέσεων από μέρους πολλών μη κυβερνητικών οργανισμών. Ευχαρίστως να σας ε, δώσω τις εκθέσεις αυτές και για αφρικανικές χώρες και στην Ασία, πώς στηρίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναπτυξιακά προγράμματα. Ευχαρίστως όλα αυτά είναι στη διάθεσή σας, αλλά δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπλουμ. Um, yes. Ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο εδώ γιατί θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να σας βοηθήσουν. Εγώ ήμουν 35 χρόνια διευθυντή σε τράπεζα στον κλάδο των επενδύσεων και πρέπει να σας πω πως δεν αγόρασα ποτέ κακή τράπεζα και δεν αγόρασα ποτέ κακό αμοιβαίο για τους πελάτες μου. Τα τελευταία χρόνια όμως πολιτικοί και οι γραφειοκράτες μου έχουν βάλει το πιστόλι στον κρόταφο και ως φορολογούμενος αγοράζω κακές τράπεζες παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε κανείς να μετρήσει στα δάχτυλα των δύο χεριών και όχι μόνο αγγλικές κακές τράπεζες αλλά ευρωπαϊκές και όλα αυτά βγαίνουν από την τσέπη του Βερτανού φορολογούμενου που έβαλε το χέρι βαθιά στην τσέπη για να στηρίξει την Πορτογαλία. Αν έχω σκοπό λοιπόν να επενδύσω ε, στο εξωτερικό θα αγοράσω αμοιβέ σε ένα-δύο αγορές. Δεν θέλω να αγοράσω μια ε, τράπεζα ε, κάκιστη και όταν λέω κάκιστη τι εννοώ η οποία έχει όλο κακά δάνεια που μάλιστα έχει εθνικοποιηθεί κιόλα. Τώρα δεν ξέρω ποιο σα συμβουλεύει, αλλά μα λέτε ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Ο καιρό δεν έχει αλλάξει εδώ και 16 χρόνια. Γιατί λοιπόν θέλετε να πετάξουμε τα λεφτά μα σε τέτοιου είδου επενδύσει. Ούτε έχω εγώ σκοπό να χάσω τα δικά μου λεφτά, ούτε οι Βρετανοί φορολογούμενοι. Και αν θέλετε να διατηρήσετε τα 3α συν, θα σα έλεγα να μην ακούσετε όσα σα λένε εδώ οι διάφοροι χαραμοφάιδε και να μην αγοράσετε τέτοιου είδους ε, τέτοιου είδους τράπεζες γιατί βέβαια αν κάνετε τέτοιου είδους ανοησίες θα χάσετε την αξιολόγηση που έχετε που είναι 3α συν. Ναι, νομίζω ότι αν ακούσει κανείς τον Βρετανό μιλητή διαπιστώνει ότι υπάρχει μεγάλη βία μεγάλη βία που έτσι και αλλιώ χαρακτηρίζει τις χρηματαγορές σήμερα. Αλλά σαφώς αν κοιτάξει κανείς τις επενδύσεις των τελευταίων ετών, βλέπει ότι τα πράγματα διακατέχονται από αυτήν την βία. Όπως είπε πραγματικά και ο κύριος Κλούτε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πραγματικά ένα εργαλείο που επηρεάζει την σημερινή ευρωπαϊκή οικονομία. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται και εκτός της Ευρώπης. Υπάρχουν σήμερα όλο και περισσότεροι Κινέζοι επενδυτές, οι οποίοι σε τρίτες χώρες χρηματοδοτούν μεγάλα έργα, μεγάλα έργα υποδομής. Πού είναι η Ευρωπαϊκή ε, τράπεζα επενδύσεων σε αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύω πραγματικά ότι εδώ πρέπει να ξαναδούμε αυτήν την πολιτική μας και βεβαίως πολύ σημαντικός τομέας που και άλλοι προανέφεραν είναι ο τομέας της ενέργειας. Ε, κοιτώντας ε, το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία θα πρέπει και εδώ να ξαναδούμε τη στρατηγική μας. Σας ευχαριστώ κύριε Μάρτιν, ο κύριος Κοζέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της ΕΤΕ, μετά από αυτά που άκουσα, που δεν είναι ε, αξιοπρεπή για, το, για αυτή την ολομέλεια, θα ήθελα να πω ότι η δράση της ΕΤΕ είναι ιδιαίτερα θετική. Οι βελτιώσεις που επέφερε η συνθήκη της Λισαβόνας δίνουν περισσότερο περιθώριο ελιγμών έτσι ώστε να δοθούν απαντήσεις στην παγκόσμια κρίση. Η ΕΤΕ, όπως υπογραμμίσατε, υποστηρίζει πραγματικά τις ΜΜΕ και συνεισφέρει στον στόχο σύγκλησης της πολιτικής για τη συνοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να συνεχιστούν και να διευρυνθούν. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις δραστηριότητα της ΕΤΕ στην Ευρώπη και θα ήθελα να υποστηρίξετε εκείνους που ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την ε, μακροχρόνια χρηματοδότηση και ιδιαίτερα ως προς τα αποταμιευτικά προγράμματα. Πιστεύω ότι η νομοθεσία περί τραπεζών και περί λογιστικής δεν λαμβάνουν υπόψη τις μακροχρόνιες επενδύσεις και τις στυλιτεύουν. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζονται μόνο προσαρμογές, χρειάζεται και μία μακροχρόνια χρηματοδότηση για να δημιουργήσουμε ένα νέο οικονομικό ορίζοντα. Έχετε δίκιο ότι η ΕΤΕ είναι μοχλός δραστηριότητας και γι' αυτό θα πρέπει να προωθηθούν δραστηριότητες ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση των χωρών της Μεσογείου. Με βάση τους κλειδονισμούς που γνωρίζουν αυτές οι χώρες, η ΕΤΕ θα μπορούσε να προβεί σε στόχοθετήσεις για την οικονομική δραστηριότητα των χωρών της Μεσογείου έτσι ώστε να προωθήσουμε τα δημοκρατικά πολιτεύματα αυτών των χωρών που έχουν αβέβαιο μέλλον. Είδα ότι είσαστε διατεθειμένος να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση μετά από αίτημα της Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Κοζέ. Ο κύριος Σάνσος Πρεζέδο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της ΕΤΕ, Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κούτας για την εξαιρετική του έκθεση. Η ΕΤΕ θα πρέπει να δράσει τάχιστα και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σε όλους τους οικονομικούς τομείς και έχει μεγαλύτερη ευθύνη τώρα κατά την περίοδο της κρίσης. Η κρίση δημιούργησε δυσκολίες εξέβρεσης πιστώσεων για να ε, σταθεροποιήσουμε το οικονομικό μας μοντέλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη φερεγγιότητα και οικονομική όρη έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κεφαλαιαγοράς και να πραγματοποιήσουμε τα κατάλληλα προγράμματα τα οποία διαφορετικά δεν θα χρηματοδοτούνταν εάν δεν υπήρχαν θετικοί όροι. Θα πρέπει το 2009 να λάβουμε υπόψη ότι η ΕΤΕ αύξησε τις ε, δραστηριότητες κατά 40% εκ των οποίων το 22% αφορά τις ΜΜΕ και την καταπολέμηση των ε, κλιματικών αλλαγών. Όμως χρειάζεται μία βιώσιμη ε, ανάπτυξη και υποστήριξη για τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση επέφερε μία επιβράδυνση αυτών των δραστηριοτήτων. Ως προς τα ευρωμόλογα θα πρέπει να εξεύρουμε νέα μέσα μέσα στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας για να φτάσουμε σε μία κοινή πλατφόρμα με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και ο εσωτερικός κανονισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις επενδύσεις της εσωτερικής αγοράς. Ο κύριος Έλες είναι ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, εγώ προσωπώ το Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω πως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να κάνουμε κάποιες θετικές αλλαγές. Ο κύριος Μπλουμ δεν εκπροσωπεί τους Βρετανούς φορολογούμενους γιατί δεν εκπροσωπείται καν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και δεν έχει καν την ελπίδα να εκλέξει ένα βουλευτή στο Κοινοβούλιο αυτό. Ας εξηγήσουμε λοιπόν τι σημαίνει ρεαλιστική πολιτική και πώς μπορεί ο φορολογούμενος με λίγους πόρους να πάρει κάτι το οποίο είναι ε, θετικό αποτέλεσμα. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ ο κύριος Μίστατ και έχει κάνει πολλά για να βελτιώσει ε, την αξιοπιστία του Ιδρύματός. Τώρα για τα ομόλογα έργου, τα project bonds, τι θα γίνει τον Ιούνιο θα παρουσιάσετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις ή έγγραφα παράλληλα με αυτά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να εισακουστείτε τη στιγμή που θα προετοιμάσετε το πολιετές πλαίσιο για την χρηματοδότηση είναι προτάσεις για ομόλογα έργου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για τις υποδομές, μεταφορές κτλ. Και τέλος, ε, τι σημαίνει αυτό, ότι θα έχουμε κάποιες οικονομίες ε, στα διαστρωτικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής, τα οποία θα μπορέσουμε τα κονδύλια να τα μεταφέρουμε και να τα κοινοποιήσουμε για τη δημιουργία αυτών των δυνατοτήτων ανάπτυξης εν ώψη της ε, στρατηγικής για το 2020. Ο κ. Μουργκάντη, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 θέτει υπόψη ορισμένους βασικούς στόχους. Θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες έτσι ώστε οι ΜΜΕ να έχουν καλύτερη προσβασιμότητα στις πιστώσεις. Επίσης τα ευρωμόλογα είναι ένα βασικό μέσο για να προωθήσουμε τον στρατηγικό τομέα των υποδομών. Όμως αμφιβάλλω για τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΤΕ, όπου χρειάζονται περισσότεροι ανθρώπινοι και ηλικοί πόροι. Το 2009 βλέπουμε πολλές δικαιούχους χώρες και βλέπω ότι η Τουρκία έχει τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με τις πιστώσεις αυτές. Λαμβάνει το 1 τρίτον και πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η Ιταλία είναι ένας από τους βασικότερους ε, μετόχους της ΜΠΕΙ και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η δυσαναλογία. Γιατί δηλαδή δίνονται τόσο μεγάλες πιστώσεις στην Τουρκία που βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόσο περιεσμένη πόλη, πόρη στην Ιταλία που τους χρειάζεται, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο κύριος Στογιάννοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ε, σπάνιο να βρεθούμε ενώπιον μία τόσο σαφούς έκθεσης. Οπωσδήποτε ο ρόλος της ΕΤΕ είναι άκρο σημαντικός. Θα ήθελα όμως να κάνω ορισμένα σχόλια ως προς την έκθεση αυτή και αυτά που άκουσα. Καταρχήν, η ΕΤΕ θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη της ΜΜΕ και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία από την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Η τράπεζα θα πρέπει να επικεντρωθεί πολύ περισσότερο σε αυτό το τομέα σε σχέση με τις πράσινες τεχνολογίες. Βεβαίω, η πράσινη τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και τις ΜΜΕ έμεσα. Σε επίπεδο Ευρώπης, εσωτερικής δηλαδή, ενδοκινοτικής πολιτικής, συμφωνώ με την άποψη Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, διότι ο έλεγχος αυτός συνάδει με τις δραστηριότητες της νέας τραπεζικής αρχής. Όμως υπάρχουν πολλές ανησυχίες και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος ως προς επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε τις ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν περισσότερα ε, κονδύλια από τις εντός. Η ΕΤΕ πάντα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με την ε, παρούσα κρίση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα την πιστοτική ε, κρίση και να δημιουργηθούν στρατηγικές υποδομές για την ανάπτυξη ολόκληρης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το σχέδιο TEN-T ε, για τις ιδιοδρομικές διασυνδέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε τις πιστώσεις και τις μικροπιστώσεις για τις υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύω ότι τα ευρωομόλογα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕ. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις ΜΜΕ και πιστεύω ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕ θα πρέπει να προβαίνει σε αυτές τις στοχοθετήσεις. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για ορισμένε δραστηριότητες της ΕΤΕ πολλές ΜΜΕ δεν έχουν επαρκή προσβασιμότητα γιατί χρειάζονται πολύ μεγάλοι πόροι. Άρα οι μικρές χώρες, οι ΜΜΕ δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ως προς τα θέματα χρόνου, πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος, στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο τομέας των ΜΜΕ. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΜΜΕ επειδή δεν σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό ιστό, θα πρέπει η ΕΤΕ να άρει αυτό το γραφειοκρατικό φόρτο. Η ΕΤΕ μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ε, ρόλο στα πρόσφατα γεγονότα στην ε, απέναντι όχθη της Μεσογείου και μπορεί να ε, υλοποιήσει μία μακροχρόνια επενδυτική πολιτική με βάση συγκεκριμένες επιλογές για την δημοκρατία και την αγορά ε, εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λούμπλιξον έχει το λόγο. Λούμπλιξον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημαντικά σημεία. Καταρχήν η ΕΤΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Αυτό σημαίνει βεβαίως και επενδύσεις για την πράσινη τεχνολογία. Για να έχουμε μια δυνατή Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, σιδηροδρομικές ε, υποδομές, τις οδικές αρτηρίες και τα λιμάνια. Οι υποδομές θα πρέπει να είναι ένα εύρυθμο πλαίσιο και η ΕΤΕ θα πρέπει να είναι πιο δραστηρία σε αυτό τον βασικό τομέα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία όταν μιλάμε για ευέλικτες οικονομικές λύσεις. Πιστεύω ότι τα ευρωμόλογα είναι ένα πολύ καλό μέσο προς την καλή, προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να έχουμε και νέα εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης. Θα πρέπει να αναπτύξουμε πρότυπα κατά τα οποία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι περιφέρειες να μπορέσουν να συμμετάσχουν πιο παραγωγικά. Η ΕΤΕ θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στις αναπτυξιακές πολιτικές και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θα πρέπει η δραστηριότητα της ΕΤΕ να είναι πλέον διαφανής και βεβαίως να συμμετέχει και η βάση περισσότερο στη λήψη αποφάσεων και να προβάλλουμε και μια εγκάρσια προσέγγιση αντιμετώπιση θεμάτων όπως η καταπολέμηση της φτώχειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούντινγκσον. Ο κύριος Στίβενσον, τέλος, για αυτό το γύρο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ένα δις ευρώ έδωσε για την, οικοδόμηση αεροτουρμπινών στο Ηνωμένο Βασίλειο και για άλλες ΑΠΕ. Αυτό λοιπόν όντως εντάσσεται στην στρατηγική για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι πως η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι αρκετά διάφανη τη στιγμή που καλείται κανείς να εξετάσει ε, την αποτελεσματικότητα αυτών των έργων. Αυτή τη στιγμή ολικό πάρκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματολογούνται με 6 δις ευρώ. Το είπε ο κύριος Μέσταρντ. Αλλά οι αιτήσει χρηματοδότηση γίνονται απλά δεκτές όταν τις υποβάλλουν τα κράτη-μέλη χωρίς να εξετάζονται σε βάθος. Αυτό δεν είναι επαρκές. Οι εταιρείε ΑΠΕ ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, λένε πως μπορούν να αποδώσουν 30% οι ανεμοτουρμπίνες αυτές, αλλά πέρσι διαπιστώσαμε πως ήταν στο 21% η απόδοσή τους, μόνο όταν είναι πάρα πολύ κρύος ο καιρός και λειτουργούν στο μέγιστο. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία μη αποδοτική επένδυση, η οποία δεν προσφέρει πλέον εκτήματα στα νοικοκυριά και τα οποία χρειάζεται ψηλή χρηματοδότηση. Αυτό είναι σκανδαλώδες και θα πρέπει η ολική ενέργεια πλέον να μην χρηματοδοτείται από την ΕΤΕ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα λοιπόν τη διαδικασία της αυθόρμητης παρέμβασης. Catch the eye. Η κυρία Μακίνες έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον James Alice για τις ε, παρατηρήσεις που έκανε σχετικά με τα σχόλια του κυρίου Μπλουμ και να πω στους συναδέλφους του Ηνωμένου Βασίλειου αν έχουν κάποιο σχόλιο ή αν διαφωνούν δεν υπάρχει λόγος να μας προσβάλλετε για να κάνετε το σχόλιο σας είπε πως είμαστε ε, κεντρικοί, ε, βαρεμένοι ε, κτλ. Εσείς σε ποια κατηγορία νίκετε αφού μας περιγράφετε έτσι. Για την ΕΤΕ να σας πω πως η Ιρλανδία ε, στην Ιρλανδία χρηματοδοτήθηκαν ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευνοήθηκαν αυτό. Αλλά πείτε μας εσείς ως πρόεδρος πόσο προσβάσιμη είναι αυτή η χρηματοδότηση. Γιατί γίνονται ανακοινώσει, ενθουσιάζονται οι μικρομεσαίες, αλλά όταν προσπαθούν να βρουν αυτή την γραμμή πιστώσεων, πολλές φορές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο έχει πρακτική επίπτωση για τις μικρομεσαίες και θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο μετά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά σκοπός ε, της χρηματοδότησης της τράπεζας είναι να υλοποιηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει υπερβολικό βάρος για τους συμμετέχοντες. Πιστεύω πραγματικά ότι η σημερινή κατάσταση σαφώς και θα πρέπει να βελτιωθεί. Εμείς ε, θεωρούμε ότι για την χρηματοδότηση 19,2 δισεκατομμυρίων που δόθηκε τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να δοθούν πολύ περισσότερες εξηγήσεις τουλάχιστον σε εμά που συμμετείχαμε και το ίδιο θα ήθελα να πω και όσον αφορά το βάρος στο κοινοτικό προϋπολογισμό και όσον αφορά τα πολύ ψηλά επιτόκια. Η τελευταία διαδικασία ελέγχου Βεβαίω και έχει πάρα πολλέ αδυναμίε. Το ελεκτικό συνέδριο και διάφορε ρυθμιστικέ αρχέ θα πρέπει να συμμετέχουν με διαφορετικό τρόπο. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι μετρήσιμα, θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα και θα πρέπει να δούμε αν και κατά πόσον τηρούνται οι κανόνες. Η πρόταση αυτή για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να εξεταστεί έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την χρησιμοποίηση και την χρηστή διαχείριση των πόρων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μπασέσκου. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κούτας για την εξαιρετική έκθεση, πολύ καλά δομημένη. Η ΕΤΕ θα πρέπει να είναι πιο επιλεκτική και να ενδιαφέρεται στα απτά αποτελέσματα. Θα πρέπει να ασχοληθεί και με τους χρηματομεσάζοντες, χρηματοδοτικούς μεσάζοντες και αυτό που έχει σημασία είναι οι στρατηγικές επενδύσεις που είναι μακροχρόνιες. Θα πρέπει μας ενδιαφέρουν οι υποδομές και η συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαίρομαι διότι η τράπεζα ασχολείται με τις, τις ε, περιφέρειες συνοχής και με τις ΜΜΕ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντιμετώπιση της κρίσης και θα πρέπει στο site να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ώστε να φαίνεται ποιες ε, περιφέρειες έχουν λάβει αυτά τα, ε, αυτά τα ποσά. Ευχαριστώ. Ενώπιν αυτής της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη Μεσόγειο, αν λάβουμε υπόψη δε και την κρίση της, ε, τη μεγάλη κρίση της Ιαπωνίας, η ΕΤΕ έχει να συνεισφέρει εμπολής. Νομίζω ότι θα πρέπει να δράσει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρώπης. Σήμερα έχουμε την κρίση της Μεσογείου και θα πρέπει να εξεύρουμε ένα νέο μέσο στο εγγύς μέλλον ένα μέσο αρρωγής, μέσω νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Εμείς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές το θέμα των Eurobonds. Πώς θα δράσετε, πώς θα, έχουν, πώς θα ορίσετε το θέμα χρονισμού και τι θα γίνει με τα υπολοιματικά ποσά που υπάρχουν. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς ε, θα εξελιχθεί και το σχέδιο Μάργκεριτ. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη στοχοθέτηση και τα θέματα χρονισμού και πώς τα ορίζετε, πώς τα ιεραρχείτε. Ο κύριος Ρουμπίξ. κύριε Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω πως η έκθεση δράση που έχει υποβληθεί για την ΕΤΕ για την περίοδο του 2009 μπορεί να γίνει δεκτή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το τι θα γίνει στο μέλλον και πρέπει να σας πω πως θα συμφωνήσω με τους περισσότερους από τους προλαλήσαντες ομιλητές. Έφτασε η ώρα να κάνουμε ε, μια αναδρομή στην στρατηγική του παρελθόντος και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Βέβαια να δούμε πώς θα αναλωθούν οι ίδιοι πόροι που αναφέρονται ε, στον ισολογισμό της τράπεζας και να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια μακροπρόθεσμη διάθεση αυτών. Ίσως με κάποια καλύτερα συστήματα εγγυήσεων ε, και πιστεύω πως θα πρέπει κάποιοι όμιλοι να, να συνεργάζονται με, τους, με τις δημόσιες αρχές, ΣΔΙΤ δηλαδή, που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις της τράπεζας. Η κυρία Ματούλα would like to take the floor. Ο κύριος Ματούλα ζήτησε. Ευχαριστώ, κύριε Πρεσέντη. Ευχαριστώ κύριε Μάιστατ, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση για βοήθεια προς ΜΜΕ και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Οι περιφέρειες σύνοχης θα πρέπει να τύχουν τις υποστήριξης της ΕΤΕ και οι δανειοδοτήσεις θα πρέπει να προωθηθούν προς τις, τους στόχους συνοχής μέσα στα πλαίσια των υποδομών και της ανάπτυξής τους. Θα πρέπει να ληφθούν κοινέ δράσεις για την συνοχή και σύγκληση από την Κομισιόν και την ΕΤΕ. Και αυτό αφορά τις μικροπιστώσεις έτσι ώστε να δημιουργηθούν θέσεις ε, εργασίας και στις αστικές περιοχές. Ως προς το, τα Jessica, Jeremy και Jaspers, αυτά τα τρία προγράμματα θα πρέπει να πούμε ότι επέτυχαν εμπολής και έτσι θα φτάσουμε σε καινοτόμα σχέδια και στο μέλλον. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κούτας για την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος, αλλά πιστεύω και τελευταίος, είναι ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση και για τα κράτη-μέλη και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχει αποδειχθεί ότι τα κράτη που έχουν μια υγιή οικονομική δομή και που μπορούν να χρηματοδοτήσουν ορθά τις επιχειρήσεις τους μπορούν να βγουν με καλύτερο τρόπο από αυτήν την οικονομική κρίση. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου το 17% των ε, επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι θέσεις απασχόλησης είναι πάρα πολλές που εξαρτώνται από αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η διευκόλυνση, η απλοποίηση των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας είναι επίσης μια στήριξη προς αυτές τις επιχειρήσεις η ανάπτυξη στις οικονομίες μας είναι απαραίτητη για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστές, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί έναντι των Αμερικανών και των Ασιατών. Χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αποτελεσματικοί και με μια αποτελεσματική δράση μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη η οποία είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε από την οικονομική κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κούν, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι όσοι ήθελαν να πάρουν το λόγο τον πήραν και σε αυτή την περίπτωση θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να μας κάνει μια περίληψη της μέχρι τώρα συζήτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Βεβαίως και θίξατε το θέμα του ελέγχου και της ρυθμιστικής αρχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της επιτήρησης, της εποπτείας και των ρυθμιστικών αρχών που θα ελέγξουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρώ ότι βεβαίως η εξαιρετική αξιολόγηση της τράπεζας αυτής είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την ίδια ώρα ξέρουμε ότι υπάρχει ένας υπερεθνικός χαρακτήρας, διακρατικός αυτή τη τράπεζα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, όπως προβλέπει και η συνθήκη. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικά βήματα, συγκεκριμένα βήματα, για να ενισχυθεί το Συμβούλιο Εποπτείας. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η τράπεζα υπάρχει η ανάγκη αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και βεβαίως το θέμα της ρυθμιστικής αρχής που θα ασκεί τον έλεγχο είναι κάτι που θα πρέπει να το λύσουμε. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να βρεθεί και μια άλλη λύση, μια εθελοντική λύση που θα βρεθεί μεταξύ όλων των ε, συμβαλόμενων μερών. Η συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν εξαιρετική και εδώ θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, παίζουμε σημαντικά ρόλο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αλλά και με την χρηματοδότηση συγκεκριμένων ε, προγραμμάτων βάσει και μέσω των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαδικασίες απαλλαγής, όπως ξέρετε, βασίζονται στις δυνατότητες που προβλέπουν τα καταστατικά και ότι ο συνδυασμός με τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την ε, υποχρεώνει να μην ακολουθεί την ίδια διαδικασία όσον αφορά την απαλλαγή. Πιστεύω πραγματικά, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια φάση μετά από την πρώτη και δυσκολότερη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι έχει τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να δοθεί νέα δυνατότητα στα καινοτόμα εργαλεία που διαθέτουμε. Θέλουμε να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση προς την έρευνα, την καινοτομία, πολύ σημαντικούς τομείς, και βεβαίως με την εμπειρία που διαθέτουμε σε αυτόν τον τομέα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καινοτόμα εργαλεία και σε άλλους τομείς εκτός της έρευνας και κοινοτομίας. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μέστατ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους πήραν το λόγο για τα σχόλια που έκαναν, ακόμα και αν κάποιοι από αυτούς ήταν λίγο, ακολούθησαν λίγο λάθος δρόμο στις σκέψεις τους. Για τον χρόνο που έχω δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις με λεπτομέρειες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά νομίζω ότι μας ζητήθηκε γενικά να κάνουμε μια πιο ενδελεχή εξέταση και κυρίως έχουμε την ερώτηση κυρίας Ιχουμπνερ. Αν θέλετε εσείς η ΕΤΕ να μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εφαρμογή και στην υλοποίηση στρατηγικής Ευρώπη 2020, μέσω της ε, σύστασης ενός κοινού μέσου εργαλείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το επιτρέπει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε υποσυζήτηση το νέο σχεδίο χρηματοδοτικού κανονισμού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσετε πως η ΕΤΕ θα είναι σε θέση να συνεισφέρει. Η πρόταση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτή την άποψη είναι κατάλληλη. Αυτό που χρειάζεται είναι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δεχτούν την πρόταση αυτή. Έχετε λοιπόν και εσείς το ρόλο που θα σας επιτρέψει να το κάνετε στο θέμα αυτό για τον χρηματοδοτικό κανονισμό. Τώρα για κάποια άλλα από τα θέματα που θίξατε, δηλαδή η φορολογική παράδειση, τα όσα είπε ο κύριος Κανφίν, Μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως η ΕΤΕ για το σημείο αυτό ακολουθεί μια πολιτική πιο αυστηρή από ό,τι άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα. Και γι' αυτό έχουμε αρνηθεί συγχρηματοδότηση με την Αφρικανική ε, Τράπεζα Ανάπτυξης ή με την Παγκόσμια Τράπεζα ή ε, και με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης χρηματοδότηση κάποιων project. Θεωρήσαμε πως αυτό δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί. Δεν πρόκειται εμείς λοιπόν να χρηματοδοτήσουμε κάποιον επενδυτή ο οποίος βρίσκεται στο μαύρο κατάλογο του ΩΣΑ. Τώρα αν θέλετε μπορώ να σα απαντήσω και με μεγαλύτερε λεπτομέρειε. Γιατί όσο είπε ο κ. Κλούτε, πιστώσεις για τις μικρομεσαίες και διαφάνεια. Δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά χρηματοστατικά όργανα που δίνουν τόσες πληροφορίες ε, για τις επιδοτήσεις για τις μικρομεσαίες και εδώ υπογραμμίζω πως ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ευνοήθηκαν από πιστώσεις που διέθεσε η ΕΤΕ έχει αυξηθεί και έχουμε φτάσει στα πάνω, στις πάνω από 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2010. Να σταθώ σε τρία στοιχεία τα οποία ε, μας έχουν κάνει μοναδικούς. Πρώτα απ' όλα, αντίθετα με τα οποία κάποια από εσά, εμείς δεν χρησιμοποιούμε το, τα χρήματα των φορολογουμένων δεν έχουμε ζητήσει ούτε ένα σέντ από τους φορολογουμένους του Ηνωμένου Βασιλείου για να στο ξεκαθαρίσω. Αυτό που χρησιμοποιούμε είναι οι πόροι που ε, ανακύπτουν κάθε μέρα από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχουμε αξιολόγηση 3α συν. Από τη ΣΥΠΑ, από την Ασία δανειζόμαστε και με αυτά που συλλέγουμε είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε υπό συνθήκες αυτά τα διάφορα έργα. Η μόνη δημοσιονομική επίπτωση είναι οι εγγυήσει για την πολιτική ρίσκου, κινδύνου δηλαδή, για την εφαρμογή της εξωτερικής εντολής που μας δίνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εκεί όντως χρησιμοποιούμε μία εγγύηση η οποία έχει κάποιο προσωρινό ε, αντίκτυπο στον προϋπολογισμό γιατί είναι το 9% των δανείων που γίνονται βασιζόμενοι στην εξωτερική διαταγή και καταπίπτει εκεί σε δύο χρόνια μετά τον πρώτη δόση του δανεισμού. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε την εγγύηση αυτή. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν χρησιμοποιείται, είναι μηδενικό το κόστος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Βλέπετε λοιπόν πως εμείς δεν κοστίζουμε τίποτα στο φορολογούμενο. Δεύτερον, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πραγματικά και μοναδικά Ευρωπαίοι. Οι μέτοχοι είναι όλα και μόνο, αποκλειστικά και μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε, έχουμε την νομική υποχρέωση μέσω των συνθήκων να στηρίξουμε οικονομικά τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είμαστε το μόνο χρηματοδοτικό ίδρυμα που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει κάποιο έργο εάν δεν λάβει προηγουμένως την θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδοτεί μετά από εξετασή που γίνεται από όλες τις γενικές διευθύνσεις. Ανταγωνισμός μέχρι περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε με αυστηρό τρόπο τις πολιτικές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ελέγχει το ελεκτικό συνέδριο. Σύμφωνα με το όσα λέει η τριμερή συμφωνία. Είμαστε σε συνεχή επαφή με την Όλαφ. Και έχουμε δεχτεί και την εποπτεία της νέας τραπεζικής αρχής, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, τουλάχιστον για την ΕΤΕ. Εμείς είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε αυτού του είδους την επίσημη εποπτεία πλέον. Το κάναμε έτσι καλώς έμεσα στο παρελθόν και κυρίως με την Επιτροπή Επαλήθευσης που έχουν εποπτική εμπειρία και το επιβεβαιώνω για μια φορά ακόμα, είμαστε απόλυτα ανοιχτοί σε τέτοιου είδους εποπτεία από τη νέα αυτή αρχή, τη νέα αυτή ευρωπαϊκή αρχή. Και το τρίτο στοιχείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ πριν κλείσω, είναι πως η ΕΤΕ είναι μοναδική στο είδος της. Γιατί έχει ε, μια διαφορετική ε, πραγματογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει. Γιατί έχουμε μόνιμο προσωπικό, πάνω από 100 μηχανικούς και επίσης εξειδικευμένους συμβούλους. Σε κάποιους κλάδους έχουμε εμπειρία και πραγματογνωμοσύνη που έχει αναγνωριστεί. Και το τεκμηριένω λέγοντας πως μας ζητούν τεχνική βοήθεια και αρρωγή για έργα τα οποία εμεί δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε γιατί γίνονται σε κάποια περιοχή που βρίσκεται εκτός της εντολής μας. Άρα λοιπόν, θα ήταν κρίμα να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την πραγματογνωμοσύνη για, τη, ας πούμε, για τις αστικές συγκοινωνίες, για την ενεργειακή ε, οικονομία, για τον κύκλο του ύδατος, για τις μικρομεσαίες. Εμείς εκεί έχουμε την εμπειρία και την πραγματογνωμοσύνη που μας κάνει μοναδικούς. Θα ήταν λοιπόν κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό σε βάθος. Και αυτό μέσα σε μια πιο συστηματική και μια πιο διαστρωμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θέσαμε ερωτήματα τα οποία νομιμοποιούνται. Εάν χρηματοδοτήσουμε, αν χρηματοδοτούμε περισσότερο στην Τουρκία είναι γιατί αυτή είναι η εντολή μας, η οποία αποφασίστηκε από κοινού, από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και μας έδωσε αυτή την αποστολή, όπου πρέπει να χρηματοδοτούμε περισσότερες υποψήφιες χώρες Δηλαδή αναλογικά ε, στην, περισσότερο στην Κροατία, στην Τουρκία από ό,τι σε άλλα κράτη. Εμείς είμαστε εκεί που είμαστε για να εφαρμόσουμε την εντολή που μας έχει δοθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές και κυρίως από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν πως αυτό δικαιολογεί μία πιο συστηματική και διαρθρωμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Τέλος, το λόγο έχει ο κύριος Κούτας, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν σε αυτή την επικοδομητική συζήτηση και θα πρέπει να αναγνωρίσω παρά ορισμένες επικρίσεις, κύριε Μαϊστάτ, ότι όλοι αναγνώρισαν το ρόλο της ΕΤΕ στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής παρούσας κρίσης. Βεβαίως χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις φιλόδοξες ιδέες. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να προβάλλουμε τέτοιες θαραλέες ιδέες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τη διαφάνεια και να υπάρχει ίσως καλύτερη επικοινωνία με όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Επίσης, εξ ονόματος των συναδέλφων, μπορώ να σας πω, κύριε το ότι μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει κλείσει η συζήτηση λοιπόν για την ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα στις 12. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερής